Ο Πρόεδρος. Ε, συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση με τις επεξηγήσεις ψήφου. Πριν περάσουμε σε αυτό, θα ήθελα να καλωσορίσω μια αντιπροσωπεία ε, του Καναδικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και ε, προσώπους τη αποστολή του Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο διπλωματικό θεωρείο. Επικεφαλή είναι ο κύριο David Τίλσον που εκπροσωπεί την εκλογική περιφέρεια του Τορόντο και συμμετέχουν βουλευτέ και γερουσιαστέ από το Κεμπέκ και τη Βρετανική Κολομβία. Έχει έρθει η αντιπροσωπή στο Στρασβούργο για να συναντήσει ομολόγου τη από την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, επ' ευκαιρία τη 34η ε, Διακοινοβουλευτική Συνέλευση ε, Καναδά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εχθές και σήμερα είχαν την ευκαιρία να ε, συναντηθούν με τα μέλη και ε, θα μεταβούν συνέχεια στη Κοπεχάγη για επαφές με την επόμενη ε, Προεδρία του Συμβουλίου. Σας καλωσορίζω και καλή διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ερχόμαστε στις επεξηγήσεις ψήφου για τις εκθέσεις που ψηφίσαμε